άξιον θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα για την Ολομέλεια. Και τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, στο σχέδιο εργασία. Το τελικό σχέδιο α, της ημερήσιας διάταξης που αποφάσισε τη σκέπτη του Προέδρου σας διανεμήθηκε για την Τρίτη. Η ομάδα του ECR σε ό,τι αφορά τη εκλογή της ε, ε, Επιτροπής, σε ό,τι αφορά την... Ε, κατάσταση στην Ιταλία και την Ελλάδα να μπει αυτό στην ε, ημερική διάταξη. Ο καθηγητή Μαριά έχει το λόγο. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του ECR ζητούμε την Τρίτη να υπάρξει δήλωση της ύπατης εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής της κυρίας Άστον για το σοβαρό θέμα της καταστροφής του χημικού οπλοστασίου της συρίας εντός της μεσογείου. αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι κάτι πολύ σοβαρό. επάνω στο πλοίο του αμερικανικού ναυτικού το cape ray γίνεται καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της συρίας με τη μέθοδο της υδρόλυσης. αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θέλουμε να συζητηθεί εδώ. η διαδικασία θα κρατήσει τουλάχιστον 60 ημέρες για τον λόγο αυτό θέλουμε να υπάρξει τοποθέτηση ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβει το συμβούλιο και η επιτροπή αν έχουν λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων σε ποιο βαθμό έχουν ενημερωθεί οι γειτονικέ περιοχές και τι πρέπει να γίνει. θέση μας είναι ότι πρέπει η καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της συρίας να γίνει εκτός της μεσογείου σε απομακρυσμένη περιοχή και ακατοίκητη ε, το εγχείρημα που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο υπάρχουν αντιδράσεις από τους πολίτες πολλών κρατών ιδίως από την κρήτη και θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό θέμα. Ε, θέλουμε λοιπόν να συζητηθεί αύριο για να υπάρξει τοποθέτηση επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένας ομιλητής υπέρ και ένας κατά της πρότασης παρακαλώ. Καταρχάς, ποιος θέλει να μιλήσει υπέρ του αιτήματο. Η κυρία Χάρμς έχει το λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Εμείς συμφωνούμε ότι το χημικό απλοστάσιο πρέπει να καταστραφεί, αλλά το θέμα της ποιότητας του, της διαδικασίας, το θέμα των περιβαλλοντικών συνεπειών, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και συμφωνεί η ομάδα μου να συζητηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Φων Στόρχ θέλει να μιλήσει κατά του αιτήματο. Α, όχι. Εντάξει, θέλει κανεί το λόγο κατά του αιτήματο. Όχι. Να ψηφίσουμε. Ποιο είναι υπέρ του αιτήματο, παρακαλώ, να σηκώσει το χέρι του. Κατά του αιτήματο. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. ηλεκτρονικό έλεγχος.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 148 υπέρ, κατά 139, 57 αποχές, εγκρίνεται το αίτημα. Και τώρα για την τρίτη υπάρχουν άλλες, ε, άλλα αιτήματα. Ja, Sie haben sich wieder gemeldet. Ist das zur Tagesordnung? ist πάλι το λόγο για την ημερήσια διάταξη. Tagesordnung für Dienstag. Μερίσια διάταξη για την Τρίτη. Bin ich zu hören? Jetzt bin ich Ναι, με ακούτε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω εγώ μια παρατήρηση να κάνω για το αυριανό θέμα Κατάλαβα ότι η προθεσμία έχει λήξει για την αλλαγή της ημερήσιας διατάξης, αλλά θα ήθελα να θέσω κάτι πολύ σύντομο και πολύ βασικό. Αύριο θα συζητήσουμε το πιο σημαντικό άτομο, την πιο σημαντική θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα πέντε χρόνια. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πιο σημαντικό αξίωμα που έχουμε να παραχωρήσουμε και έχουμε 90 λεπτά χρόνο ομιλίας. Όπως ε, και στην, ε, το χρόνο που ε, χρειαστήκαμε για να συζητήσουμε τα περί για παράδειγμα. Θεωρώ ότι η σημαντικότητα, η σημασία του θέματος το οποίο συζητάμε αύριο δεν ελήφθη υπόψη και θα πρέπει να σεβαστούμε τον πολίτη. Δεν είναι δυνατόν 90 λεπτά μόνο να έχουμε να συζητήσουμε και μία πρόταση για το πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Όχι, όχι, όχι λέει ο Πρόεδρος, αυτό είναι θέμα διαδικαστικό. Δεν είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περνάμε τώρα στην Τετάρτη λέει ο Πρόεδρος. Εδώ η ομάδα της ΓΚΟΕ σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης ζητήθηκε ψήφισμα. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρίες και κύριοι, η κυρία Καβιτσίμερ. Θα ήθελα εξ στην ομάδα μου να ζητήσω την Τετάρτη το απόγευμα όχι μόνο να υπάρξει ομιλία και συζητήσει σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, αλλά να υπάρξει και ψήφισμα, να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα, γιατί η κατάσταση ε, κλιμακώθηκε περαιτέρω το Σαββατοκυριακό και ω Κοινοβούλιο ε, θα τα πούμε και θα συνεδριάσουμε μετά τις θερινέ διακοπέ. Είναι λοιπόν κατεπήγον να ε, εκφραστούμε όχι μόνο να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με την ε, είπατε εκπρόσωπο, αλλά να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποτραπεί περαιτέρω βία. Πάνω από 170 είναι νεκροί, ε, εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ισραήλ και χιλιάδες ε, Παλαιστίνοι φεύγουν, αναγκάζονται να φύγουν από το βόρειο τμήμα της ε, Γάζας, απειλούνται και επαπειλείται επίθεση εδάφους. Θα πρέπει λοιπόν θεωρούμε σαφώς να τοποθετηθεί το κοινοβούλιο μας. Υπέρ του αιτήματο, ο, ο κύριος Γκερερό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, δεν θα πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας για την κλιμάκωση της βίας στην περιοχή αυτή. Θα πρέπει από τώρα να στείλουμε ένα μήνυμα ώστε οι εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν μια αυτοσυγκράτηση και να καταπαύσουν το πυρ. Είμαστε υπέρ ενός ψηφίσματος και αν καταφέρουμε να εκφράσουμε στο ψήφισμά μα, τη στεναρή και ενωμένη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα στηρίξει τις προσπάθειες άλλων παραγόντων για να ε, σταματήσει η βία θα ήταν πολύ θετικό. Θα θέλαμε ένα σύντομο ψήφισμα που θα ζητά κατάπαυση του πυρός, θερματισμό ε, της βίας και από τις δύο πλευρές, επαναφορά του διαλόγου και σεβασμό όλων των κατοίκων της περιοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς να μιλήσει κατά του αιτήματο αυτού. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε υπέρ της διεξαγωγής συζήτηση, αλλά κατά της σύνταξης ψηφίσματος. Πολύ αμφιβάλλω αν είναι σκόπιμο να συντάξουμε ένα σύντομο ψήφισμα και με ένα σύντομο ψήφισμα να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ, μέσα σε δύο μέρες και όλα, ή όπως ζήτησαν οι σοσιαλιστές. Πολύ αμφιβάλλω κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, το αίτημα, λοιπόν, είναι ε, δηλώσεις με ψήφισμα. Να το ψηφίσουμε, λοιπόν. Όποιος συμφωνεί με την αίτηση της ε, ΓΚΟΕ, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Ποιος είναι κατά του αιτήματο αυτού. Άποχες. Σαφής πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι λοιπόν ε, ορίζεται και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα εργασίας για την τρέχουσα εβδομάδα. Και περνάμε λοιπόν τώρα στις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού. Πρώτος ο ομιλητής, ο κύριος Τσακάη. Έχετε το λόγο. Herr Τσακάη. Ja, bitte sehr. Okay. Thank you, Mr. President.